ότι χειρεύει πλέον η έδρα της από 14 Δεκεμβρίου 2010 και μετά κατόπιν. Η ομάδα ε, των Δημοκρατών και Φιλελευθέρων μου ζήτησαν ε, να διορίσω τον κύριο Γιωχάνες Κορνέλης Φανμπάλεν στην διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν θα αντικαταστήσει τον κύριο Καρλ Χάγκλουντ. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Οπότε εγκρίνεται ο διορισμός του. Αλλαγές στην ημερήσια διάταξη τώρα.